Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο από τις 9 μέχρι τις 1 και από τις 3 ε, μέχρι τις 5. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λύεται η συνεδρίαση.